Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στη συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών. Κυρίσω την έναρξη των εργασιών μας. Πριν ξεκινήσω όμως, ε, ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μια αντιπροσωπεία μας μετέβη την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα και θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την αξιέπαινη προσπάθειά της, κυρίως την Έμιλη και το Ράντεκ, γιατί ήταν τόσο άρτη η διοργάνωση με τέτοιο υψηλό επαγγελματισμό και τόσο ε, απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών που πραγματικά αξίζουν χειροκρότημα οι υπάλληλοι της γραμματείας, γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολη η προετοιμασία αυτή της περίπλοκης αποστολής. Και νομίζω ότι νιώσαμε ιδιαίτερη περηφάνεια τα μέλη της αντιπροσωπείας ε, και πραγματικά αναγνώρισαν και είναι ε, για την άρτια προσπάθειά σας και την άμεμπτη διοργάνωση αυτής της αποστολής. Βιμ, καλή σου μέρα! Ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Ήταν μια πολύ αποτελεσματική αποστολή αυτή, πολύ ενημερωτική και η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, έτσι δεν περιμένει εμά καθόλου. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και στον τομέα των μεταφορών, τι συμβαίνει στην Κίνα. Υπάρχει όμως ε, και μία μικρή επίκριση που θέλω να κάνω. Ε, η πτήση από το Ταϊλίν ως το Τσιντζέν είχε καθυστέρηση 2,5 ώρες. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κοιμηθήκαμε πάρα πολύ αργά. Ίσως την επόμενη φορά θα πρέπει να διορθώσουμε λίγο την κατάσταση με τις πτήσεις. Oui, mais sauf que je le ε, ναι. Αλλά γι' αυτό δεν ευθύνεται η γραμματεία για το αν θα ανοίξουν δηλαδή Κινέζοι και θέρες στις πτήσεις. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την ε, παρατήρηση που δεν μας αφορούσε και πολύ. Εν πάση περιπτώσει. Και ο κύριος Πίτερ ήταν παρόν. Πάντως ε, σίγουρα η αποστολή αυτή μα εμπλούτησε τις γνώσεις μας, ε, μας έμαθε πάρα πολλά, οπότε γίναμε πιο πλούσιοι και από διανοητική άποψη, αλλά και από ανθρώπινη άποψη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια μας διάταξη, παρακαλώ. Κύριε Άντερσεν. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που το λέω από την αρχή. Δεν είδα τα πρακτικά ακόμη, αλλά έχω ένα διαδικαστικό πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες ολομέλειας για τα δικαιώματα των επιβατών σε διεροδρομικών μεταφορών ε, και το πώς διαχειριστήκαμε την, ε, τον κατάλογο ψηφοφορίας ε, στο σχετικό θέμα. Ήταν πολύ δύσκολο το θέμα και για τη γραμματεία, το αναγνωρίζω, γιατί ήταν ε, πολύ επίμαχο το θέμα και ήταν πολύ δύσκολη η σύνταξη, η κατάρτιση του καταλόγου ψηφοφορίας. Ήταν πολύ περίπλοκος και μάλιστα έγιναν πολύ σημαντικές αλλαγές ε, χωρίς να ενημερωθούν εγκαίρως οι σκιώδεις ηγητές. Δηλαδή, μόνο τελευταία στιγμή ενημερώθηκαν για τις σημαντικές αλλαγές και παρόλο που τρει έλεγε η προθεσμία για την υποβολή σχολείων για τον κατάλογο ψηφοφορία, μπορούσαμε να επικαλεστούμε την εξαίρεση τη ανωτέρα βία. Ζήτησε το ΕΛΚ ξεχωριστή ψηφοφορία. Έχει απόλυτο δικαίωμα να το κάνει και το αποδέχομαι και μάλιστα το ζήτησαν και εμπρόθεσμα πριν την εκπνοή τη προθεσμία. Παρόλα αυτά δεν ενημερώθηκε κανεί γιατί η γραμματεία περίμενε το σύνολο του καταλόγου και εμεί συζήτηση άλλου θέματο στη συνεδρίαση των συντονιστών. Πάντως, όταν κάτι τόσο σημαντικό ανακύπτει και κοινοποιείται, θα πρέπει να ενημερώνονται όλοι σε προκαταρκτικό στάδιο και όχι την τελευταία στιγμή, δηλαδή μετά τις συνεδρίες των συντονιστών. Εγώ απουσίαζα, αλλά όταν έλαβα τις ψήφους και είδα τις ψήφους, γιατί ψηφίσαμε αμέσω μετά την επομένη το πρωί, πολλοί δεν είχαν συνειδητοποιήσει για τι ε, ρηξικέλευτε αλλαγέ που είχαν γίνει στι συμβαστικέ τροπολογίε. Ξέρω πόσο δύσκολη ήταν η θέση τη Γραμματεία σε τέτοια περίπτωση με τόσο περίπλοκο ζήτημα, αλλά ελπίζω να αποτραπεί στο παρελθόν μια επανάληψη τέτοια κατάσταση. Ευχαριστούμε κυρία Άντερσεν για τι παρατηρήσει. Καλώ τι σημειώνουμε. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Το σημειώνουμε, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω. Περνάμε τώρα στη συζήτηση του πρώτου σημείου, την πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 9653 του Συμβουλίου για την προθεσμία ε, για την εφαρμογή των ειδικών κανόνων σε ό,τι αφορά το μέγιστο μήκο στην περίπτωση θαλάμων οδήγηση που παρουσιάζουν βελτιωμένα αποτελέσματα ω προ την αεροδυναμική απόδοση, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τι επιδόσει ασφαλεία δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, δηλαδή στην υποφαινόμενη. Η οδηγία αυτή προβλέπει για κάποια οχήματα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και για τις εθνικές και για τις διεθνείς μεταφορές, καθώς και τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη για τις διεθνείς μεταφορές. Το κείμενο αυτό έχει διπλή εμβέλεια και αντίκτυπο και οικολογικό, περιβαλλοντικό, αλλά και ένα σκέλος που αφορά την ασφάλεια. Οπότε η βελτίωση της αεροδυναμικής κατάστασης των θαλάμων οδήγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων επιτρέπει σημαντικά ωφέλη για την ενεργειακή απόδοση των οχημάτων. Βέβαια, λόγω των περιορισμών που επέβαλε η Οδηγία 96-53, για, τη, τα μέγισ, για τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος ήταν αδύνατο να γίνει η μείωση χωρίς να περιοριστεί το ωφέλιμο βάρος, το ωφέλιμο φορτίο των οχημάτων. Οπότε, τι έγινε. Τροποποιήθηκε η οδηγία 96 96-53 προκειμένου να βελτιωθεί ε, η αεροδυναμική κατάσταση αυτών των μηχανοκίνητων οχημάτων και η οδική ασφάλεια, επιτρέποντας μια παρέκκληση από τις διατάξεις για το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκο, υπό κάποιε προποθέσει όμω. Παρ' όλα αυτά, τι είχαμε στο κείμενο τη τροποποίηση, με το άρθρο 9α, παράγραφο 3 τη οδηγία 719, 719, που ε, τροποποιήθηκε από την οδηγία του 2015 και που προβλέπει ένα δικαιοστάσιο, μία αναστολή τριών ετών για την θέση σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την επιμήκυση των θαλάμων οδήγησης όπως περιλαμβάνοντα, στην τελική συμβαστική λύση μεταξύ των δύο σκελών της νομοθετικής αρχής. Δεδομένη τη τρέχουσα κατάσταση και λαμβανομένου υπόψη ότι οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από τι οδικέ μεταφορέ αντιπροσωπεύουν το 1 τέταρτο των συνολικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. 1 τέταρτο, ε, δηλαδή πολύ σημαντικό μερίδιο των συνολικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιπλέον, λαμβάνοντα υπόψη οι εκπομπέ από ε, τι οδικέ μεταφορέ προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 6% στο χρονικό διάστημα 2015-2030, η Επιτροπή έκρινε ότι ε, θα πρέπει να αποσύρουμε, να ε, επωφεληθούμε το συντομότερο δυνατό από τα ωφέλη των επιμήκων θαλαμών οδήγησης. Οπότε η σημασία του θέματο αυτό επιβεβαιώνεται και από την πρόταση για τα πρότυπα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα των βαρέων φορτηγών οχημάτων που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της δέσμης μέτρων 3 για την κινητικότητα. Πράγματι, για τη συμμόρφωση με τα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα βαριά φορτηγά οχήματα θα απαιτηθεί σήμερα η εφαρμογή διαφόρων τεχνολογιών για τη βελτίωση τη ενεργειακή του απόδοση. Μεταξύ αυτών, ε, προβλέπεται και η εισαγωγή αεροδυναμικών θαλάμων οδήγησης, που είναι το αποτελεσματικότερο μέτρο για τη μείωση της οπισθέλκουσας, της αντίστασης του αέρα. Τώρα, να δούμε αυτό το θέμα της ε, τριετούς αναστολής του δικαιοστασίου. Γιατί η οδηγία που προβλέπει την αναστολή κατά τρία έτη για την εισαγωγή των αεροδυναμικών ε, θαλάμων οδήγησης από την ημερομηνία μεταφοράς η εφαρμογή των αναγκαίων τροποποιήσεων όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου. Η οδηγία αυτή λοιπόν προτάθηκε να προσαρμόσει το άρθρο 9α παράγραφος 3 ώστε να καταργηθεί η αναστολή των τριών ετών και να προβλεφθεί συντομότερη αλλά αναλογική προθεσμία. Τέλος, ε, ποιες είναι οι προτάσεις της εισηγήτριας. Ε, ήρθε επιτέλους η ώρα να συγκεκριμενοποιηθούν τα ωφέλη που αναμένονται από τους αεροδυναμικούς θαλάμους οδήγησης λόγω των ενεργειακών επιδόσεων των βαρέων φορτηγών οχημάτων αλλά και λόγω της καλύτερης ορατότητας για τους οδηγούς της ασφάλειας των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου καθώς και της ασφάλεια και της άνεσης των οδηγών. Είναι αναγκαίο λοιπόν να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η εισαγωγή αυτών των, θαλάμων, των αεροδυναμικών θαλάμων οδήγηση χωρίς περιττή καθυστέρηση. Ως εκ τούτου σας προτείνω να εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τροποποίησης. Και να την εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατό για να μεταφερθεί η οδηγία στα κράτη-μέλη με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι γίνεται σήμερα. Αυτή είναι η έκθεση και να δώσω το λόγο στους και ηγητές τώρα για τη συζήτηση, ξεκινώντας. Καλημέρα σας κύριε Μαρινέσκου. Φτάσατε καλά, έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την ε, διεξοδική παρουσίαση όπου μας εκθέσατε τα πλεονεκτήματα της πρότασης. Δεν προτείνετε τροπολογίε. Θέλετε να κρατήσετε την πρόταση της Κομισιόν αυτούσια. Αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω μία τροπολογία σήμερα για να παρατείνουμε λιγάκι την περίοδο ούτω ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Είχαμε κάποιες συζητήσει Οι 8 μήνες είναι μία πρόταση που θα γίνει αποδεκτή σχεδόν από όλου. Γι' αυτό λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε προβλήματα για τον ανταγωνισμό. Υπάρχει μια... Υπήρχε μια μακρά περίοδο που ήξεραν ήδη ότι θα υπάρξουν αυτές οι αλλαγές, επομένως η αυτοκινητοβιομηχανία προετοιμάστηκε. <clears throat> Αλλά και για να μην ακούσουμε σχόλια και παράπονα από μέρους τους, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προτείνουμε 8 μήνες. Ευχαριστώ κύριο Σασίς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με απόλυτα με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και συμφωνούμε απόλυτα και με τη δική σας πρόταση, κυρία Συγήτρια. Γιατί υπάρχουν ε, λόγια εύλογοι και οικολογικοί και ασφάλειας, ώστε να εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό αυτές τις τροποποιήσεις της οδηγίας. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα, όπως σας είπα, με τις προτάσεις της εισηγήτριας με την έκθεση λοιπόν κυρία Πρόεδρε. Και έτσι θα ψηφίσουμε. Θα υπερψηφίσουμε την πρότασή σας δηλαδή. Ευχαριστούμε κυρία Σύς. Ensuite, Monsieur Lundgren, la parole est à vous. Well, I don't δεν έχω πολλά να προσθέσω. Όλα όσα είπατε είναι σωστά. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμων και βεβαίως ε, με, την, με τους θαλάμους οδήγησης θα μειώσουμε και την αντίσταση του αέρα. Δεν πρόκειται να παρουσιάσω τροπολογίες, μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, εκτός και αν υπάρξουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις. κυρία Μέσνερ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για αυτήν την πρόταση. Δεν νομίζω ότι είναι επίμαχο το θέμα αυτό όσον αφορά την ε, εφαρμογή του λέμε ότι αυτές οι άλλες ε, καμπίνες, οι άλλοι θάλαμοι οδήγησης όχι μόνο αυξάνουν την ασφάλεια, αλλά και από οικολογικής πλευράς, όπως είπε και η κυρία εισηγήτρια, είναι πιο επιθυμητές, διότι είναι πιο αεροδυναμικές. Είχε υποθεί ότι θα πρέπει πρώτα να ε, κάνουμε δοκιμές με τις καμπίνες αυτές ε, και να έχουμε ε, μια τριετή αναστολή της εφαρμογής. Το θέμα λοιπόν είναι να τις χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αλλά το θέμα εδώ είναι τα μεγάλα φορτηγά, το μήκος τους. Νομίζω ότι ε, τα ε, φορτηγά μεγάλου μήκους ε, μπορεί να είναι πιο οικολογικά και σε κάποια κράτη-μέλη επιτρέπεται η χρήση τους, ε, δεν επιτρέπεται όμως να περάσουν τα σύνορα. Ε, έτσι λοιπόν υπάρχει εδώ μια γκρίζα ζώνη. Τι γίνεται σε περίπτωση που ε, δύο κράτη-μέλη που συνορεύουν μεταξύ τους επιτρέψουν και τα δύο αυτά τα φόρτηγα. Δεν νομίζω ότι θα εξεταστεί το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία, διότι υπήρχε επιθυμία εξέταση τη κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε το σχέδιο ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το θέμα αυτό όμω ε, συνδέεται ακριβώ με τι διαστάσει των φορτηγών και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μέσνερ. Η Κομισιόν, η κυρία Βέρνερ έχει το λόγο, πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε και κυρία Εισηγήτρια, μπορώ να είμαι πολύ σύντομη στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές για την ε, υποστήριξή τους για την ε, πρόταση αυτή. Δηλαδή, ε, προτείνουν η υιοθέτηση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την χρήση αυτών των αεροδυναμικών θαλάμων οδήγησης που εξασφαλίζουν και καλύτερη ορατότητα για τους οδηγούς και καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Λόγω της ευαισθησίας του θέματος των διαστάσεων υποβάλαμε μία ε, πολύ περιορισμένου πεδίου πρόταση για να αποφύγουμε το μορατόριο, για να μην κολλήσουμε ε, σε πολύπλοκες συζητήσεις. Εξετάζουμε ε, τους νέους ε, κανόνες έγκρισης τύπου. Οι κατασκευαστές ε, λοιπόν θα εφαρμόσουν θα ενημερωθούν ταυτόχρονα ώστε να μην έχει κάποιος ε, άδικο πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους. Πάντως πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο να ε, εφαρμοστεί η πρόταση αυτή το συντομότερο δυνατό. Θα επανέλθω στην κυρία Μάισνερ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη νομοθετική πρόταση. Εσείς αναφέρεστε ιδιαίτερα στο θέμα ε, της διέλευσης των συνόρων ε, μεταξύ δύο κρατών μελών ε, που συμφωνούν ως προς τη χρήση των μεγάλων φορτηγών. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Βέρνερ, θα απαντήσω στους συναδέλφους. Κύριε Μαρινέσκου, η περίοδος που προβλέπετε... Α, θέλετε κυρία Μάισνερ ξανά το λόγο. Ήθελα να προσθέσω το εξή. Καταρχά, ήθελα διευκρίνηση σχετικά με τη διέλευση των, των συνόρων, αλλά ο κύριος Καραμίτσος υποσχέθηκε να υποβάλει νέα πρόταση αφού εξετάσει τις εμπειρίες των διαφόρων κρατών μελών με τα μεγάλα φορτηγά. Θα είναι χρήσιμο λοιπόν να επιτρέπεται η χρήση του ευρωπαϊκού δρόμου εφόσον όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν. Προφανώ δεν φταίτε εσεί, ε, αλλά αυτά που μα υποσχέθηκε ο κύριο Καραμίτσο, πού είναι. Ερώτηση λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Μάιστα. Να απαντήσω τώρα και εγώ με τη σειρά μου για την ε, περίοδο των 8 μηνών του πρότεινε ο κύριο Μαρινέσκου. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Μπορούμε να το σκεφτούμε όμω. Εγώ θέλω να σα πω το εξή όμω. Κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμοστεί μπορούμε να διαπραγματευτούμε τους 8 ε, μήνες, αλλά 8 μήνες θα είναι το μέγιστο, δεν θα δώσουμε παραπάνω από 8 μήνες. Ε, και θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως να το ξανά συζητήσουμε το θέμα αυτό ξανά. Δεύτερον, για να απαντήσω στην κυρία Μάισνερ. Καταλαβαίνω τα ερωτηματικά σας, κυρίως για τα μεγάλα φορτηγά, τα πολύ, τα πολύ ογκώδη φορτηγά τα μεγαφορτηγά, που δεν μου αρέσει η λέξη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια γρήγορη εφαρμογή ε, και θα έπρεπε αυτά τα μεγάλα φορτηγά να μην τα εισάγουμε σε αυτό το κείμενο. Θα έπρεπε ένα άλλο κείμενο να έχουμε για αυτά. Γιατί αν περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε για να καλύψουμε και τα μεγάλα φορτηγά, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε καλύτερα. Εγώ θέλω, προτιμώ μια γρήγορη υιοθέτηση του κειμένου και έστω η επόμενη θητεία, το επόμενο κοινοβούλιο δηλαδή, να το εξετάσει. Ε, πάντως, στην, στο μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε, δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα των μεγάλων φορτηγών. Ε, 20 Νοεμβρίου είναι η προθεσμή για την κατάθεση των τροπολογιών μέχρι το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε με την πρόταση κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλίας ε, και τους δημοσιονομικούς κανόνες για τα λόγω ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και μετανάστευση, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων. Ο κύριος Ζλωτόφσκι έχει το λόγο, αλλά δεν είναι εδώ. Ποιος τον αντικαθιστά? Α, ο κύριος Ζλωτόφσκι θα έρθει όπου να είναι. Θα τον περιμένουμε λοιπόν. Ή μάλλον δεν θα τον περιμένουμε. Θα πάμε στο επόμενο σημείο. Ούτε ο επόμενο εισηγητή είναι εδώ όμω. Οπότε τι να κάνουμε, θα περιμένουμε τον κύριο, τον κύριο Είναι ήδη μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου και φτάνει όπου να είναι. Μια μικρή αναμονή.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 Allez, on peut reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Παρακαλώ. Κύριε Ζωτόφσκι, καθίστε παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ. Μια και μπήκατε. Θα σας δώσω το λόγο για να παρουσιάσετε την έκθεσή σας και εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στους ε, σκιώδες εισηγητές στην Κομισιόν και θα σας ξαναδώσω στο τέλος το λόγο, κύριε και Έχετε το λόγο για την αρχική παρουσίαση. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε για την καθυστέρηση, αλλά με καθυστέρησε η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις Βρυξέλλες. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμότατα τους και ηγητές ε, από όλες τις πολιτικές ομάδες για την πολύ ενεργό συμμετοχή τους στην κατάρτιση της γνωμοδότησής μας. 158 ε, ήταν οι τροπολογίες που καταθέσαμε στο σχέδιο της ε, Επιτροπής, κάτι που προϋποθέτει πολύ έντατη σημαντική προσπάθεια. Συμφωνώ απόλυτα με πολλές τροπολογίες και σας ευχαριστώ που τις καταθέσατε γιατί έτσι ενισχύσετε το κείμενο προκειμένου να εκφράσουμε τη θέση της Επιτροπής για τις κοινέ διατάξεις του νέου πακέτου για τα διάφορα ταμεία. Επίσης, είχαμε και κάποιες προτάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τι αρμοδιότητε τη Επιτροπής Μεταφορών. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαφωνώ με τις τροπολογίες, απλώς είναι εκτό θέματο. Καλύτερα λοιπόν να τι ε, υποβάλουμε ξεχωριστά σε ψηφοφορία μετά τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε. Κατά την κατάρτιση των συμβαστικών τροπολογιών επικεντρώθηκα κυρίω στα κέρια πιο νευραλγικά σημεία που αφαιρούν άμεσα τι επενδύσει τη μεταφορέ και άφησα κάποιες άλλες τροπολογίες εκτός του πεδίου των συμβαστικών τροπολογιών. Ε, δεν σας κρύβω ότι δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσουμε το άρθρο 104 και από τεχνική και από ουσιαστική άποψη για την κατανομή των ε, κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής. Ε, Καταρχήν ε, υπάρχουν πολλές διαφορές ε, ε μεταξύ μας ό,τι αφορά την κατανομή των κονδυλίων των εθνικών φακέλων στα 70 και 30%. Πάντως ελπίζω να καταλήξουμε σε κοινή θέση των Επιτροπών Τρακέιτρε για τα, το μηχανισμό συνδέοντα στην Ευρώπη. Και ελπίζω να έχουμε κοινή προσέγγιση των δύο επιτροπών για τα θέματα αυτά. Ε, προτιμώ βέβαια μία συγκεκριμένη θέση, αλλά θέλω να καταλήξουμε σε κοινή αποδοχή συμβαστικέ τροπολογίε ώστε να εκφράσουμε την άποψη τη Επιτροπή Μεταφορών. Ελπίζω τελικά να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για το άρθρο 104 και προσβλέπω σε καρποφόρες ε, ε, λύσεις ε, και για το άρθρο 84. Ε, θέλω ε, να σας υποβάλω εγκαίρως τις συμβαστικές τροπολογίες για να έχετε χρόνο να τις μελετήσετε και προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία με όλους. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Κύριε Ζωτόφσκι. Θα ξεκινήσουμε με τους κοιόδης συζητητές. Η κυρία Κλόντια Σμιτ ε, εκπροσωπείται από τον κύριο Βιν Βαντεν Κάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το απόγευμα έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να αντικαθιστώ την Κλάουντια Σμιτ, η οποία επιστρέφει από αποστολή. Είναι ακόμα σε ταξίδι δηλαδή. Επομένως την αντικαθιστώ σήμερα, έτσι. Ευχαριστώ Κοσμά Ζωτόφσκι για την ε, παρουσίασή σου και για το ότι μας παρουσίασε στο μήλο της έρηδας. Προσπαθούμε να καθορίσουμε ε, στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου το νέο ε, μέσο συνδέοντας για την Ευρώπη. Συνδέοντας την Ευρώπη, Και έχουμε και τα περιφερειακά ταμεία. Υπάρχει μια έκθεση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά την κατανομή, την αποτελεσματική κατανομή των δημοσιονομικών πόρων μεταξύ των ταμείων. Και συμφωνούμε ότι τα ταμεία και οι πόροι του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη, του ΣΕΦ δηλαδή, θα πρέπει να πάνε στις χώρες συνοχής. Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βάλει μια νέα ρήτρα για, την, για τον ανταγωνισμό. Ο Κοσμάς το είπε, το θέμα του 70% και του 30%. Στη δική μας ομάδα υπάρχει επίσης, πρέπει να σας το πω ειλικρινά, μια κάποια διαίρεση, έτσι, μια ρήξη για τις διάφορες αποχρώσεις των επιμέρους σημείων και θέλω να δω τι συμβιβασμός θα προκύψει ε, χάρη στις προσπάθειες του Κοσμά. Τα ταμεία συνοχής θα πρέπει να δίνουν πόρους στις χώρες συνοχής. Και διερωτώ με αν η ρήτρα με βάση τον ανταγωνισμό είναι κατάλληλη για την κατανομή των κονδυλίων. Ε, επίσης υπάρχει περιορισμός για χρησιμοποίηση των κονδυλίων για τρία χρόνια. Αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή μέσα τρία χρόνια επιστρέφουν στα ταμεία. Αυτό μου φαίνεται καλύτερο από το, τη ρήτρα του ανταγωνισμού. Ε, η Κλάουντια λέει στην Τραν, ε, λέει μάλλον η ίδια, ε, ότι συμπαθεί περισσότερο τη ρήτρα της ανταγωνιστικότητας. Σε πάση περιπτώσει, πρέπει να προσπαθήσουμε για να βρούμε ένα συμβιβασμό. Η Επιτροπή Τραν θα πρέπει να βρει το συμβασμό. Γιατί αν αφήσουμε το θέμα στη Ρέτζη ή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών θα είμαστε πολύ πιο Ευάλωτη και δεν νομίζω ότι θα βρούμε τελική λύση εύκολα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ασή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη συζήτηση για το θέμα αυτό πριν από μερικές εβδομάδες ήδη σα παρουσίασα κάποια βασικά σημεία της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που θα θέλαμε να τροποποιηθούν στην αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Γι' αυτό και καταθέσαμε και τροπολογίε προκειμένου να υλοποιήσουμε του στόχου μα. Καταρχήν, να προωθήσουμε μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών και για το, τα, τους σπόρους ε, για τις α, ε, διάφορες ε, για τις διάφορες δράσεις και η περικοπή κατά 45% του κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής είναι απαράδεκτο, απαράδεκτη και θα πρέπει να διαφωνήσουμε. Επίσης, διαφωνούμε με την ε, πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 30% των πόρων που, μετα... που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχή στο Σιδέτο στην Ευρώπη να διατίθεται σε ανταγωνιστική βάση. Επίση, ε, το ποσοστό χρηματοδότηση ε, μειώνεται και αυτό θα πλήξει τι επενδύσει στις λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχές ό,τι αφορά την υποβολή σχεδίων, ιδιαίτερα για τι μεταφορέ που θα έχουν αποφασιστική σημασία για την ανάπτυξη αυτών των περιφερειών. Επίσης θα πρέπει οι στόχοι της, των ταμείων να ευθυγραμμιστούν με την προώθηση της δίκαιης και οικονομίας και της περιφαλλοντικής, λαμβάνοντας υπόψη και τη Συμφωνία των Παρισίων. Επίσης, ε, θα θέλαμε να εφαρμόζονται με ε, με απόφαση ε, της ειδικής πλειοψηφίας ε, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, με την αντίστροφη, είναι υπέρ της αντίστροφης ε, ενισχυμένης πλειοψηφίας. Διαφωνούμε με αυτό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη δυνατότητα αναστολή τη χορήγηση κονδυλίων για χώρε που παραβιάζουν το κράτο ε, δικαίου. Ιδιαίτερα όταν παραβιάζονται κατάφορα οι αρχέ του κράτου δικαίου που αποτελούν θεμελιώδει αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ σημαντική αρχή και δεν συμφωνούμε με μια απλή εξαίρεση σε περίπτωση μη τήρηση των οικονομικών αρχών. Καταρχήν, η οι πρώτε αρχέ εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ισχύουν πολλοί παράγοντες και όχι μόνο μια πολιτική επιλογή των κρατών μελών. πέραν των τροπολογιών των άλλων συναδέλφων και πιστεύω ότι χάρη στη συνεργασία των σχεδόν εισηγητών θα καταλήξουμε σε πολλές συμβαστικές προτάσεις, όπως είπε και ο συντάκτης γνωμοδότης, προκειμένου να στηρίξουμε όλους αυτούς τους στόχους. Είμαστε εν γνώση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των ε, ομάδων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πιθανότητα αναστολή ε, τη της κονδυλίων για παραβίαση του κράτου δικαίου, αλλά πιστεύω ότι με τη συζήτηση θα προλιάνουμε το έδαφος και ελπίζω να μα στηρίξουν και άλλες πολιτικές ομάδες στη συζήτηση των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σύς. Ο κύριος Χικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. η πρόταση το να μεταφέρουμε δηλαδή λεφτά προς τον μηχανισμό ΣΕΦ είναι λογική για μια επιτροπή μεταφορών. Επίσης, μια και τα θέματα αυτά είναι λίγο γενικόλογα. Αυτό το γλίστριμα του 8% των κονδυλίων του ΦΕΝΤΕΡ προς άμεση διαχείριση ε, προς το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη είναι λογικό. Γιατί το, ο μηχανισμός αυτός το ΣΕΦ δεν έχει αρκετά λεφτά. Και είχαμε διάφορους διαγωνισμούς όπου η προσφορά ήταν μεγαλύτερη από την ζήτηση. Και επίσης θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τα δίκτυα TNT που χρειάζονται 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν έχουμε. Επομένω, το πρώτο θέμα είναι ε, τα ποσοστά και η κατανομή των κονδυλίων. Θα το πρέπει να το συζητήσουμε με τον εισηγητή φυσικά, με την εισηγήτρια. Η Επιτροπή Μεταφορών θεωρεί ότι καλύτερα θα ήταν να υπάρχει άμεση διαχείριση των χρημάτων ε, και να δοθούν εκεί που υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενα αξία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο. Υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στρέφομαι τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκυγιόμ, αλλά ξέχασα τον κύριο Μαρινέσκου, οπότε πρώτα ο κύριος Μαρινέσκου. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να επανέλθω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το 75%. Αυτή τη στιγμή στην διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, στην πρόταση αυτή, όσον αφορά τις μεταφορές, η πρόταση είναι να διατηρήσουμε το ισχύον ποσοστό ε, να μειώσουμε όμως ε, το χρονικό διάστημα στα δύο χρόνια. Επί δύο χρόνια λοιπόν κάθε κράτος μέλος θα χρησιμοποιεί ε, την, ε, τους πόρους από την πολιτική συνοχής και μετά το πέρασμα των δύο αυτών ετών νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη συμβιβαστική λύση. Ε, τα χρήματα που δεν θα έχουν απορροφηθεί να χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη ε, σε ανταγωνιστική βάση. Και έτσι θα λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση των περιφερειών στο κάθε κράτος μέλος και η δυνατότητα των κρατών μελών για να δαπανίσουν τους πόρους αυτούς για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, διότι ξέρετε ότι ε, οι πόροι αυτοί προσωπηθούν μόνο για τις μεταφορές και για το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, με την πρότασή μας ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πλαίσιο προγραμμάτων, μάλλον ένα πρόγραμμα πλαίσιο διορθώνει ο μιλητής. Νομίζω ότι έτσι τα κράτη-μέλη θα είναι καλύτερα σε θέση να υποβάλουν κάποια καλά προγράμματα. Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω τον εισηγητή να εξετάσει τις ε, τροπολογίες μου, διότι στη γνωμοδότηση δεν προκύπτει σαφώς ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα χρηματοδοτεί μόνο προγράμματα περιβάλλοντος και μεταφορών. Σας ευχαριστώ. Merci Ευχαριστούμε. Κύριε Μαρινέσκου, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιλόντ, ο κύριος Βίμ Βαντενκάμπ θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, κυρία, κυρία Πρόεδρε, έχω κάποιες παρατηρήσεις εδώ της Κλάουντια Σμιτ που είναι σκιώδης εισηγήτρια για ε, το ΕΛ. θα ήθελα όμως να πάρω το λόγο και στο όνομα του Ντίτερ Κοχ ιδιαίτερα όσον αφορά την τροπολογία 35 που είναι δική του και έχει να κάνει με την ασφάλεια στον τομέα των μεταφορών. Θα ήθελα λοιπόν στο όνομα του Ντίτερ Κόχ να ρωτήσω τον κόσμο Σλοτόφσκι Θα ήθελα να τον παρακαλέσω να εξετάσει ιδιαίτερα αυτήν την τροπολογία 35, που είναι του Ντίτερ Κόχ και έχει να κάνει με την ασφάλεια στις μεταφορές. Σας ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις ε, εκ μέρους κάποιου άλλου μέλους του ΕΛΚ ή η ευρωπαικη Επιτροπή του Λόγου. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο σήμερα. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αναγνώριση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλούστευση ε, της πολιτικής συνοχής και πιο εύκολη πρόσβαση στους πόρους, καθώς και για αναγνώριση της ισορροπίας που έχουμε πετύχει όσον αφορά τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους από τη μία και την προστασία ε, ε, της νομιμότητας των δαπανών. Επιτρέψτε μου να απαντήσω πολύ σύντομα, διότι έγιναν κάποιες παρατηρήσεις ε, σχετικά με τα χαμηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού. Το θέμα αυτό συνδέεται με την διασφάλιση του γενικότερου της γενικότερη δέσμης επενδύσεων. Όσο πιο ε, υψηλό το ποσοστό χρηματοδότηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο ε, πιο περιορισμένη θα είναι η τελική πόρη. Θέλουμε εμεί όμω να μεγιστοποιήσουμε τις επενδύσεις σε όλη την πολιτική συνοχή και στις μεταφορές. Λαμβάνω γνώση των όσων υπόθηκαν ε, σχετικά με τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη και θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον εισηγητή ε, στις προσπάθειες επίτευξης συμβιβασμού δεδομένης της διαφορετικής κατεύθυνσης που ακολουθούν οι διάφορες τροπολογίες. Δεν θα σας εκπλήσει ότι κατά τη γνώμη μα η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ισορροπημένη και ε, διατηρεί το επίπεδο μεταφοράς πόρων που είχαμε για το διάστημα 2014-2019. Θεωρούμε όμως ότι αυξημένοι πόροι στην αρχή του διαστήματος αυτού θα επιτρέψουν πιο γρήγορη χρηματοδότηση προγραμμάτων που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν και έτσι θα έχουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο κύριος Μαρινέσκου τόνισε το θέμα του Ταμείου Συνοχής ε, και της ε, εστίασης ε, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Το Ταμείο αυτό όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα πράγματα επίσης, διότι το πεδίο εφαρμογή του είναι πιο ευρύ και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατά της μεταφοράς πόρων από την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Και τέλος, ε, μια παρατήρηση για το κράτος δικαίου που αναφέρθηκε επανειλημμένα εδώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στο θέμα αυτό, καταρχάς επειδή δεν εμπίπτει στι αρμοδιότητες μου, αλλά και επειδή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού αυτού, υπάρχει μερική αναφορά σε μια αιτιολογική σκέψη σχετικά με ξεχωριστή πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα κράτου δικαίου. Ε, δεν θα πρέπει αυτό το θέμα να το χειριστούμε στην τομεακή νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ξανά ο εισηγητή έχει το λόγο για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Πολύ σύντομα. Θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη όλες σας τις παρατηρήσεις και τις τροπολογίες που αναφέρονται στην καλύτερη λειτουργικότητα του συστήματος μεταφορών και θέλουν να τη βελτιώσουν. Ενώ άλλε τροπολογίες θα τι αφήσουν να ψηφιστούν ξεχωριστά. Τώρα για την τροπολογία περιθμό 35 του κυρίου Κοχ θα της αφιερώσω ιδιαίτερη προσοχή όπως μου ζητήσατε και να τονίσω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση του κυρίου Μαρινέσκου. Και αυτή θα πρέπει να την εξετάσουμε και να τη λάβουμε υπόψη σε κάποιο βαθμό. Αυτά. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζομαι τις συμβαστικές τροπολογίες και θα τις υποβάλω στον Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ζωτόφσκι. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου, όπως προβλέπετε. Συνεχίζουμε με την έκθεση που αφορά την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές παροχής υπηρεσιών από λεωφορεία και πούλμαν. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ρόμπερτ Τζίλε. Ευχαριστώ, Καρίμα. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η σημασία των μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και οι κοινοί κανόνες για την πρόσβαση στη διεθνή αγορά τέτοιου είδου ε, υπηρεσία είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα γιατί αφορά πολλούς συμπολίτε μας που χρησιμοποιούν τέτοιες μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν και υπάρχει και πολιτικός αντίκτυπος ε, αυτής της κατάστασης έξω και οι 370 τροπολογίες που έχουμε λάβει για την έκθεσή μου. Δεν μας εκπλήσει αυτό, ούτε μας ευνηδιάζει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και είναι πολλά θέματα που θέλουμε να συμφωλιώσουμε. Τα χώρισα σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη ομάδα, στην πρώτη κατηγορία, είναι οι συνάδελφοι που θέλουν να κρατήσουν τις εθνικές αγορές παροχής υπηρεσιών με λεωφορεία και πούλμαν σχεδόν απολύτως κλειστές. Η δεύτερη ομάδα των συναδέλφων έχουν κάποιε επιφυλάξει ω προ την θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ω προ τη δική μου που είναι κάπως πιο ήπια και θέλησε να βρει κάποιε συμβαστικέ προτάσει και υπάρχει και μια τρίτη ομάδα συναδέλφων που δεν ακούγεται και πολύ ε, και που είναι περισσότερο υπέρ της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τάσσονταν υπέρ ακόμη και μεγαλύτερης απελευθέρωσης αυτής της αγοράς. Θα σταθώ λοιπόν στα πιο κεντρικά θέματα που προσπαθούμε να να συμφωνήσουμε με τους και ηγητές. Το πιο καθόδες θέμα είναι αυτής οι υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών, PSO, PSO. Και υπάρχουν τρεις ομάδες υφερόντων γύρω από τις συμβαστικές τροπολογίες. Είχαμε όμως πολλές συζητήσεις και με τους ε, συμφεροντούχους από τις αγορές και τις επιχειρήσεις που και αυτές είναι διχασμένες. Ε, υπάρχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορα κράτη-μέλη, αλλά και ε, τα Υπουργεία Μεταφορών θα ήθελαν να κρατήσουν τις υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών ως έχουν, σε εθνικό επίπεδο δηλαδή. Αυτό κράτησα από τις άριθμες συναντήσεις που είχαμε. Πάντω πιστεύω ότι για τι ε, υποχρεώσει παροχή δημοσίων υπηρεσιών μπορούμε να καταλήξουμε σε πιο ελαστικέ προτάσει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να μην τις καταστρέψουν αυτές οι υποχρεώσεις εκεί που λειτουργούν, αλλά ε, καλό θα είναι σε μερικές περιπτώσεις να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Τώρα για τους θερματικούς σταθμούς. Και εκεί, μετά από κάποιες συζητήσεις που είχαμε τους και ηγητές, αρχίζουμε και κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, διαχωρίζουμε τους ε, ορισμούς των τερματικών σταθμών από τους ορισμούς για τους επιβάτες και δεν κολλάμε σε θέματα εμβαδού ή παροχή υπηρεσιών όπως αποχωρητήρια και το καθεξής. Ε, το εντάσσουμε στα πλαίσια της συγκεκριμένης νομοθεσίας στο θέμα των τερματικών σταθμών. Και σε θέμα των εθνικών αδειών ε, ισχύουν οι κανόνες σε κάθε κράτος μέλος και δεν ε, πάδουμε από αυτούς. τώρα, οι ρυθμιστικές αρχές Πιστεύω θα καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις, αν και ακόμη υπάρχει διάσταση απόψεων. Θέλω να κρατήσω τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι επαφείται στα κράτη-μέλη να συστήσουν αυτές τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές. Δεν μπορεί πάντως να είναι η ίδια νομική οντότητα η ρυθμιστική αρχή και η αρχή που οργανώνει του τους δημόσιους για τις κρατικές προμήθειες, για τις δημόσιες συμβάσεις. Θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός για να έχουμε καλή λύση. Για το καμποτάζ μεταφορές και αυτό είναι ακαθόδες θέμα. Δεν μπορούμε για άλλα θέματα να έχουμε καλό καμποτάζ και για, ε, κακό καμποτάζ και για τα λεωφορεία και πούλμα να είναι καλές οι ενδομεταφορές. Για τις υπόλοιπες μεταφορές ε, αγαθών να είναι κακό το καμποτάζ για μεταφορές Τώρα, θα πρέπει να γίνεται εύκολη η καταχώρηση ε, μία επιχείρηση αν θέλει να δραστηριοποιηθεί σε άλλη αγορά. Αν γίνεται όμω αμέσω δεν μιλάμε καν για καμποτάζ. Μερικές φορές όμως αναβάλλεται κατά ένα εξάμεινο η έναρξη λειτουργία μια επιχείρηση Οπότε σε τέτοια περίπτωση μα ενδιαφέρει το θέμα του καμποτάζ. Αν δεν γίνει άμεση εφαρμογή τη ε, άμεση θέση σε λειτουργία τη επιχείρηση. Πάντω, είχαμε πολλές συναντήσει ήδη με τους σκιώδει ηγητέ και προβλέπονται αρκετέ ακόμη, γιατί μετά την τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Στρασβούργο διαπιστώσαμε κάποια καθυστέρηση στη διαδικασία. 13 Νοεμβρίου θα έχουμε την επόμενη συνεδρία στο των σκιωδών εισηγητών ε, και προτείνω η ψηφοφορία να γίνει 22 Ιανουαρίου, κάπως αργότερα από ό,τι προβλεπόταν αρχικά, γιατί θα έχουμε και το Δεκέμβριο συνεδριάσει των σκιωδών εισηγητών, ώστε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ τους και οδησηγητές. Ελπίζω να συνεχίσουμε την επικοδομητική συνεργασία και να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Ζήλε. Ο κύριος Βιμ Βαντενκάμπ δικαστήριο τον κύριο Ντεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ο κύριος Ντεγκράντες Δυστυχώ έχει μία συνεδρίαση εκτό της Επιτροπής Μεταφορών και δεν είναι διαθέσιμος ε, σήμερα το απόγευμα. Ε, η απόψη του είναι η εξή. Θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την κατανόηση που δείχνει για τις δυσκολίες που συνδέονται με αυτή την έκθεση και για την ε, θέλησή του να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Όπως ακούσατε και στην εισαγωγή του κ. Ζήλα, είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο. Τρεις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών έχουν γίνει και στην τελευταία συνάντηση ο εισηγητής παρουσίασε 20 συμβαστικές τροπολογίες. Η βασική ιδέα, οι βασικές ιδέες θέλουμε να εκφραστούν. Ο κύριος de ε, grandes Μα είπε ότι συζητήθηκαν διάφορα θέματα μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και προσπαθούν να, βρουν συμβασμού για τα βασικά θέματα. Καταρχά, ε, το κανονιστικό ρυθμιστικό όργανο, ε, καθώ και ποιο αποφασίζει για την ε, άδεια για τα 100 χιλιόμετρα. το βασικό θέμα αυτό συνδέεται με το άρθρο 8. Οι διαδικασίες δηλαδή αδειοδότησης για τις διεθνείς μεταφορές. Όπως ξέρετε, η πρόταση της Κομισιόν μιλούσε για κάποια όρια για τις ε, εθνικές αγορές, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει με διαφορετικό τρόπο τα κράτη-μέλη και η δυσκολία είναι ακριβώς αυτό το επίπεδο. Οι συγητές θα πρέπει να βρουν συνένεση σε ό,τι αφορά τα σημεία που πρέπει να λάβουν τα σημεία μάλλον που συνδέονται με τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Αυτό το σχέδιο καονισμού είναι μια απόπειρα απάντησης ε, στις ανάγκες της ενιαίας αγοράς για την οποία παλέψαμε. Ε, θα πρέπει να επιτευχθούν οι συμβιβασμοί ούτως ώστε να έχουμε πιο φιλελεύθερη, πιο ασφαλή και πιο δίκαιο οικονομικό σύστημα. Ε, οι δρόμοι είναι ραχοκοκαλιά της Ευρώπης και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και είναι ο πιο κοινωνικό δίκαιος μέσω, ε, τρόπος μεταφορών. Στις 22 ε, Ιανουαρίου λοιπόν θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών. Έχουμε λοιπόν χρόνο, θεωρούμε, θεωρούν οι εισηγητές, αλλά μην ξεχνάτε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πρέπει να το προσέξουμε πραγματικά. Εκ μέρου του κυρίου Ντεγκράντε ευχαριστώ όλου που κατέθεσαν τροπολογίε. Είναι ανοιχτό και αυτό για να συνεχίσει να συζητάει, ούτω ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Βαντενκάμπ. Η κυρία Άντερσον θα πάρει το λόγο και θα ε, προσωπήσει τον κύριο Κόβατσεφ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόβατσεκ ζητεί συγγνώμη που έπρεπε να αποχωρήσει διότι είναι πλήρες μέλος της Ήτρε και έπρεπε οπωσδήποτε να βρίσκεται εκεί. Όσον αφορά τις απόψεις του, πιστεύει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι όσον αφορά τις ε, εθνικές και διεθνείς μεταφορές ε, επιβατών, πέρα από τον κανονισμό 1073 και και τον ε, κανονισμό για τις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια στη νομοθεσία αυτή και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό προτείνει προσέγγιση με εξαίρεση της εφαρμογής ε, αυτού του κανονισμού, διότι έχει να κάνει με την ελευθέρωση τη εσωτερική αγοράς και πιστεύει ότι θα υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους δύο κανονισμούς. Και άλλοι το έχουν αναφέρει αυτό στις ε, διάφορες τροπολογίες. Προτείνει λοιπόν ε, στον εισηγητή να ζητηθεί γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δέχεται ελευθέρωση του τομέα των πούλμαν και των λεωφορείων. Επίσης, ε, προτείνει ευέλικτη προσέγγιση στις τροπολογίες του να ε, ε, εναπόκειται στα κράτη-μέλη το αν θα ελευθερωθεί η αγορά ή όχι. Το κατόφλι των 100 χιλιόμετρων δεν αντιστοιχεί στις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τη διαρθρωτική δομή. Θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να μπορεί να θέτει μόνο του το κατόφλι και πολλά μέλη του S&D συμφωνούν μαζί, συμφωνούν μαζί του. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης ε, για το κόστος ε, μη κερδοφόρων γραμμών είτε με τέλη είτε με κρατικές ενισχύσεις. Επίσης έχει εξετάσει τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι και που ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση. Θα ε, ήθελε να παρακαλέσει τον εισηγητή τις προτάσεις να τις ομαδοποιήσει σε τρεις ε, κατηγορίες. Ε, ελευθέρωση, καθόλου ελευθέρωση και διάμεση λύση. Ε, αυτή η προσέγγιση νομίζω ότι είναι επικοδομητική όσον αφορά την εξέβριση συμβασμού και χαίρομαι που ακούω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Επίσης, όσον αφορά την δημιουργία νέου οργανισμού, ε, οι εργασίες αυτές στα περισσότερα κράτη-μέλη πραγματοποιούνται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε ένα νέο ε, ρυθμιστικό σώμα με υψηλό κόστος λειτουργίας. Συμφωνεί λοιπόν ότι αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα, ε, χωρίς ε, όμως ε, να έχουμε επιπλέον κόστος. Γνωρίζετε τις απόψεις του για τις ενδομεταφορές και όσον αφορά τις μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων. Πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και όσον αφορά τους θερματικούς σταθμούς διαφωνεί όσον αφορά το εμβαδόν ε, και βλέπει ότι στις τροπολογίες ότι αρκετοί συνάδελφοι συμφωνούν μαζί του. Δεν έχει ασχοληθεί περαιτέρω με το θέμα των ε, τερματικών σταθμών. Πιστεύει όμω ότι πρέπει να στηρίξουμε τη συνάδελφο Λούση Άντερσον, παραθέτω τα λόγια του, ε, όσον αφορά του οικονομικού φορεί και τι σχετικέ απαιτήσει. Και λαμβάνω γνώση και των τροπολογιών Σελίτσκα και στο θέμα αυτό. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί υπεραιτέρω ε, σε, τι, σε ποιο στάδιο προβλέπεται η καταχώρηση των ε, λεωφορείων στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Merci beaucoup, Madame Anderson. Ευχαριστούμε, κύριε Άντερσον. Κυρία Ουλκοπ. Ουσκοπα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που άργησα. Χαίρομαι όμως που ε, μπόρεσα να είμαι παρόν τελικά και θα μιλήσω σχετικά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νομοθεσία που αφορά ε, εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς λεωφορείων σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό καθήκον για μας να φροντίσουμε οι συνθήκες εργασίας των οδηγών λεωφορείων να είναι όσο γίνεται ε, καλύτερες και να λαμβάνουν και δίκαιη αμοιβή που να ανταποκρίνεται στις διαδρομές που οδηγούν. Θα πρέπει επίσης ε, να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ε, υψηλό επίπεδο ασφαλείας στις οδικές μεταφορές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια καλή αγορά στον τομέα αυτών στην Ευρώπη ε, και να μην μειώσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, πιστεύω, να Υπάρχει πρόσωπο από την επιχείρηση των μεταφορών στην χώρα όπου πραγματοποιούνται οι μεταφορές και να μπορούν οι αρμόδιες αρχές ε, να ε, διαπιστώνουν ε, εάν τηρούνται οι κανόνες. Έχουμε δει τρομερά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια. Είδαμε πολλούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες και αυτό ακριβώς υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής νομοθετικής ρύθμισης στον τομέα αυτών. Επίσης, είναι σημαντικό οι ενδομεταφορές ε, να ε, πραγματοποιούνται ε, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιούνται και οι μεταφορές εμπορευμάτων οι ενδομεταφορές εμπορευμάτων. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Είναι κεντρικό για την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης. Την ευχαριστώ και που ήρθε. Ξέχασα τον κύριο Ρικέ. Τον ξέχασα. Ζητώ συγγνώμη κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Για τη δουλειά διαμεσολάβησης που έκανε για ένα λεπτό θέμα όπου υπάρχουν διαφορετικές θέσεις λόγω των ε, εθνικών παραδόσεων. Εκεί όπου οι μεταφορές ε, με λεωφορεία και πούλμαν είναι βασικό στοιχείο των δημοσίων μεταφορών και οργανώνεται σε αυτά τα πλαίσια, υπάρχουν μεγάλες αντιστάσεις για οποιαδήποτε αλλαγή του ισχύοντος συστήματος. Ενώ όταν μειώνεται ο ρόλος των δημοσίων μεταφορών υπάρχει σε αυτές τις χώρες μια μεγαλύτερη δυνατότητα ανοίγματο. Η θέση του εισηγητή είναι μια θέση ισορροπίας. Ε, με μεγάλη δεξιότητα μας ε, οδήγησε ως εδώ. Για τη δική μας ε, ομάδα, τέσσερα-πέντε στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν θα επανέλθω στο θέμα των ε, των δημοσίων, της παροχής δημοσίων υπηρεσιών είναι μια ε, αένα ή μια τέρμονη συζήτηση αυτή. Τα, με, όσοι είναι υπέρ του μονοπωλίου του δημοσίου θέλουν, ε, βάζουν πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις για αυτές τις ε, συμβάσεις ε, δημοσίων υπηρεσιών. Θα πρέπει να δούμε ε, τι ισορροπία θα βρούμε ανάμεσα αυτήν την υποχρέωση παροχής δημοσίων υπηρεσιών και στο άνοιγμα. Εκεί όπου συμφωνώ με τον εισηγητή είναι ότι ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες ε, θα πρέπει να δούμε τι ορισμό θα έχουμε στους τερματικούς σταθμούς. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τις παραδόσεις που έχουμε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να αφήσουμε κάποιο περιθώριο ελιγμών σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε απλούς ορισμούς, λειτουργικούς ορισμούς, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να μπορούν να δώσουν ε, διευκρινήσεις. Τώρα, για τις ρυθμίσεις. Ε, πολλοί μίλησαν άσχημα. Ορισμένοι είπαν ότι είναι διοικητικό άχθος. Αλλά στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ανοίγματο στην αγορά, που το θέλουν οι αν δεν υπάρχει ρυθμιστικό όργανο, νέο, ανεξάρτητο, δεσμευτικό, δεν υπάρχει πιο άνοιγμα. Η ιδέα λοιπόν ότι τα ρυθμιστικά όργανα των δημοσίων προμηθειών αυτοί που ρυθμίζουν δηλαδή τις ε, δημόσιες συμβάσει ε, είναι και ρυθμιστικά όργανα, δεν είναι σωστό. Πρέπει να τα δείτε όλα αυτά και να δείτε τι συνέβη στου ε, ε Εάν δεν υπάρχει υποχρεωτικό τέτοιο όργανο, ρυθμιστικό όργανο, δεν υπάρχει άνοιγμα. Ε, εάν είμαστε κατά του ανοίγματο, στην πραγματικότητα θέλουμε να καταργήσουμε το ρυθμιστικό όργανο για τις διαδικασίε αδειοδότηση, να λάβουμε υπόψη τι παραδόσει των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να υποχρεώσουμε να δοθούν άδειε ανοιχτέ παντού, ε, ειδικά σε κρατημέλη που έχουν πολύ σημαντικού σημαντικές οδικές μεταφορές. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο το έργο του εισηγητή. Ε, θα πρέπει όμως και να προστατεύσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, εκεί όπου είναι πολύ σημαντικές και ανεπτυγμένες, ε, καλά διαρθρωμένες, χωρίς όμως να καταδικάσουμε το πνεύμα του καονισμού, που είναι δηλαδή το πνεύμα του ανοίγματο. Θέλουμε οι ενδομεταφορές να ληφθούν υπόψη, δεν μπορούμε να τις αφήσουμε εκτός. Επίσης, ε, η συνάδελφος μόλις μίλησε για το καμποτάζ. Όταν το αντιμετωπίσουμε άσχημα, ε, βαρύνει ολόκληρο τον κανονισμό. Σε αυτή την περίπτωση, ένα καλό κείμενο για τις συνθήκες εγκατάστασης που λαμβάνει υπόψη και τις ενδομεταφορές για τις ε, μεταφορές προσώπων θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε τα προβλήματα και τα λάθη που διαπράξαμε για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Είναι δύσκολη αυτή η νομοθεσία, λεπτή. Φυσικά θέλουμε να υπάρξει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και άρα άνοιγμα, γιατί αυτό ακριβώς ε, πλαισιώνει την Ευρώπη και οι οδικές μεταφορές ε, επιβατών βεβαίως είναι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όπως όλες οι υπόλοιπε μεταφορές ε, οδικού τύπου. Φυσικά η... δεν θα πρέπει ή τα τομεακά συμφέροντα των διαφόρων κρατών μελών να αποδυναμώσουν αυτή την ε, πρόταση που είναι το τελευταίο πρόβλημα ε, που πρέπει να ρυθμίσουμε για τις μεταφορές γενικά. Ούτως ώστε να έχουμε και στον τομέα των οδικών μεταφορών επιβατών ε, ένα σύστημα μεταφορών που αξίζει και προσυδειάζει στον 21ο αιώνα. Να μην έχουμε δηλαδή οδικές μεταφορές όλων των υπολείπων πραγμάτων του 21ου αιώνα και των επιβατών του 20ου αιώνα. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε τη θέση της Κομισιόν. Η κυρία Βέρνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζήλε για τις συνεχείς προσπάθειες του προκειμένου να βρεθεί ισορροπία στο θέμα αυτό. Εκτιμούμε ιδιαίτερως ε, την προσπάθειά σας να καταλήξετε στις συμβαστικές ε, τροπολογίες, συνδυάζοντα τις τροπολογίες των συναδέλφων σας. Όπως είπατε κι εσείς, ε, έχουμε τρεις ομάδες θεμάτων στις οποίες θα ήθελα να σταθούμε. Τα βασικά θέματα αφορούν την προστασία των συμβάσεων, των δημοσίων συμβάσεων, κοινοφελών υπηρεσιών ή τη υποχρέωση παροχή δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να βρεθεί ισορροπία μεταξύ των θεμετών συμφερόντων των μεταφορέων που έχουν ε, συμβάσει ε, δημοσίων υπηρεσιών και των αρμοδίων αρχών με τις αρμόδιες εργασίες και να το συμφιλιώσουμε με την ανάγκη ενός ε, στιβαρού κανονιστικού πλαισίου για, την παροχή υπηρεσιών μεταφορών με πουλμαν και λεωφορεία, ώστε να δρέψουμε τα ωφέλη, ε, τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά από τις μεταφορές αυτές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το μέσο δρόμο, τη χρυσή τομή, για να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των ε, συγκρόμενων αυτών στόχων. Δηλαδή να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να απορρίψουν εμπορικέ υπηρεσίε που μπορούν να διαταράξουν την οικονομική ισορροπία τέτοιων δημοσίων συμβάσεων. Και επίση προβλέπουμε τροπολογίε, ώστε να έχουμε περιορισμένη χρήση αν ε, μπορεί να εξεταστεί εναλλακτικό δρομολόγιο. Σε ό,τι αφορά το, τις ενδομεταφορές και την πρόσβαση στην αγορά. Και εδώ η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από την κατάσταση που έχουμε στις μεταφορές εμπορευμάτων. Εκεί έχουμε προγραμματισμένες υπηρεσίες και αξιοσιοδοτημένες που επίσης μπορούν να ελεγχθούν. Υπάρχει και εδώ δυνατότητα να βρούμε τη σωστή λύση χάρη στο κριτήριο της εγκατάστασης και στο κριτήριο της πρόσβασης της αγοράς και μάλιστα σε μια συνδυασμένη εφαρμογή τους. Δεύτερη σημαντική ομάδα θεμάτων αφορά τους τερματικούς σταθμούς. Πολλές τροπολογίες προτείνουν τη χρήση του ορισμού του τερματικού σταθμού που παρέχεται στην οδηγία και τον κανονισμό 181 του 2011 για τα δικαιώματα των επιβατών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί όμως ότι η πρόσβαση για πρόσβαση χωρίς διακρίση υπηρεσίες συλλοφορίων και πουλμάν θα πρέπει να ισχύει για περισσότερους θερματικούς σταθμού από αυτού που αναφέρονται στον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών, γιατί υπάρχουν εμ, περιορισμοί σε θέματα προσωπικού και εγκαταστάσεων και ε, περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό τερματικών σταθμών ε, με βάση το πώς το εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Δεν είναι κατά τη γνώμη μας σωστός ορισμός για να επιτρέψουμε εξάπλωση τέτοιων υπηρεσιών πουλμαν και λεωφορείων. Και τελευταία ομάδα θεμάτων ε, αφορά τα κανονιστικά σώματα, τους κανονιστικούς φορείς, ρυθμιστικούς φορείς. Έχουμε μεγάλες ανησυχίες ε, γιατί κάποιες τροπολογίες προσπαθούν να αποδυναμώσουν το ρόλο των ρυθμιστικών φορέων. Κατά τη γνώμη μας ε, προέχει να είναι ο ρυθμιστικός φορέας ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο για να χαίρει εμπιστοσύνη και θα θέλαμε οι αποφάσει του να λαμβάνονται με αντικειμενικό τρόπο σε μια αναφιόμενη αγορά, χωρί μεροληψίε και χωρί σύγκρουση συμφερόντων. Κάτι που θα ίσχυε αν ήταν η αρμόδια αρχή και για την περίπτωση της ε, των συμβάσεων. Επίση όπω έχουμε και στις σιδεροδρομικέ μεταφορέ, θέλουμε ένα εξάρτητο ρυθμιστικό φορέα. Πολύ συχνά, σε πολλά κρατημέλη, είναι ίδιος ο ρυθμιστικός φορέας που έχει αρμοδιότητα για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και για τις υπηρεσίες λεωφορείων και πούλμαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βέρνερ. Ο κύριος Ζήλ έχει το λόγο για να ολοκληρώσουμε. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ Καρίμα, ευχαριστώ τους συναδέλφου που ζήτησαν το λόγο και υπέβαλαν παρατηρήσεις. Ξέχασα δύο θέματα στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Στη συναντήρηση των σχεδόν εισηγητών είπαμε ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί ο ορισμός και να μιλήσουμε για ε, συγκεκριμένες μεταφορές μεταξύ των ε, πόλων για και πούλμαν. Επίσης, σε μερικές ε, χώρες έχουμε μονοπωλιακή κατάσταση στις αγορές αυτές. Έχουμε λοιπόν κάποια ιδιαίτερα δικαιώματα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που θα πρέπει να προσέξουν την κατάσταση τη μονοπωλιακή. Και έχουμε ε, ρυθμιστικές αρχές όχι μόνο στις οδικές μεταφορές αλλά και σε άλλους κλάδους και δεν είναι τόσο δαπανηρή αυτή η λύση. Και μέσω και μακροπρόθεσμα θα μας εξασφαλίσει ε, ποιοτικέ υπηρεσίε σε προσιτέ τιμέ ε, για του πελάτε που είναι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε τέτοια προσέγγιση και για τις υπηρεσίες ε, από λεωφορεία και πούλμαν. Και εξακολουθεί να είναι σχετικά κλειστός αυτός ο τομέας των μεταφορών ακόμη. Και ίσως θα ήταν από τα τελευταία, από τους τελευταίους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί, ενώ οι τηλεπικοινωνίες ή άλλοι ε, τομείς έχουν ε, απελευθερωθεί πολύ πιο νωρίς. Φανταστείτε, αν και για την καινοτομία υιοθετούσαμε τόσο κλειστή προσέγγιση, ε, πώς θα προχωρούσαμε στα θέματα του Ευρωπαϊκού εθέρα, για παράδειγμα. Σίγουρα με τον ανταγωνισμό έχουμε μετά από μερικά χρόνια πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι με τα μονοπόλια και από άποψη κόστου και από άποψη ποιότητα ε, των υπηρεσιών που παρέχονται, ο ανταγωνισμό κατά τη γνώμη μου, είναι η καλύτερη λύση. Πιστεύω ότι με του και ηγητέ ε, και με την παράταση του χρονοδιαγράμματο θα καταφέρουμε να καταλήξουμε στι συμβαστικέ προτάσει. Ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά. Να σα υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή θα γίνει στι 22 Ιανουαρίου του 2019. Και συνεχίζουμε με την επόμενη μας έκθεση που αφορά την οδηγία για τις δράσεις εκπροσώπησης των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την οδηγία 2009-22. Δυστυχώς απουσιάζει ο κύριος Μάιερ, ο εισηγητής μας, οπότε δύσκολο είναι να έχουμε συζήτηση ερήμην του εισηγητού του συντάκτου της γνωμοδότησης. Και μάλιστα δεν έχει και δικαιολογήσει την απουσία του ο κύριος Μάγερ, ο συντάκτης γνωμοδότησης. Τι θα γίνει, προχωρήσουμε στη συζήτηση. Αν είναι παρόντε και και θέλουν να σχολιάσουν έστω και την απουσία του συντάκτη γνωμοδότηση, ε, έχουν την ευκαιρία. Κύριε Βίμ Κάμπ, θέλετε να Μιλήσετε εκ μέρους του κυρίου Μαρινέσκου. Όχι, από τους σοσιαλιστές επίσης. Απουσιάζει ο συντάκτης γνωμοδότησης. Πάντως η ψηφοφορία θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου. Δεν έχει νόημα να δώσουμε το λόγο ούτε στον κύριο Μπορκ, μια και απουσιάζει ο συντάκτης γνωμοδότησης. Μα λείπει ο συντάκτη γνωμοδότηση. ο εισηγητή απουσιάζει. Οπότε ε, υπάρχουν τουλάχιστον βοηθοί για να κρατήσουν σημειώσει από τη συζήτηση. για να μπορέσει να λάβει υπόψη της ε, τα σχόλια που θα, ακούσει στη συζήτηση, που θα ακουστούν στη συζήτηση. Αν δεν υπάρχει κάποιο να κρατάει σημειώσει για να ενημερώσει τον ε, εισηγητή αργότερα, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε. Δυστυχώς δεν πληρώνονται οι προϋποθέσεις. Οπότε δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να σας ενημερώσω απλώς ότι η ψηφοφορία μας θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου και ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε άλλη συνεδρίαση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών. Λυπάμαι, αλλά δεν Φταίω εγώ αν ε, εμφανίζεται ή αν επουσιάζει κάποιος συζητητής. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που προβλέπουν ε, τη σύσταση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ναυτιλιακής θηρίδας με βάση την οδηγία 2010-65. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κλούν, η κυρια κλουνα επίσης απουσιάζει. Donc, je vais faire une pause de 5 minutes. Οπότε θα έλεγα να διακόψουμε για ένα πεντάλεπτο. Γιατί μου είπαν ότι θα την αντικαταστήσει ο κύριος Βιμ Καμπ. Οπότε διακόπτουμε για 8 λεπτά. Voilà. Je... Hein? Yes, is, is she, is...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

Allez, nous allons Συνεχίζουμε. Ξαναρχίζουμε τις εργασίες, παρακαλώ. Παρακαλώ, ας συγκεντρωθούμε. Η κυρία Κλούν είναι εδώ. Έχουμε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει ένα σύστημα ενίας ευρωπαϊκής θηρίδας. Κάντε πολύ θόρυβο. Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Θηρίδα που θα, ε, θα καταργήσει την ε, οδηγία του 2010, την 65. Ε, Κυρία Κλούν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν για μια ευρωπαϊκή ενιαία ναυτιλιακή θηρίδα. Γιατί θα είναι και υπέρ του ανταγωνισμού και τη αποτελεσματικότητα του ναυτιλιακού τομέα. Θα πρέπει να μειώσουμε το διοικητικό άχθο για τα πλοία και να χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή θα πρέπει να... Ε, κάθε φορά που ελμενίζεται ένα πλοίο και ελμενίζεται κάθε χρόνο, κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια πλοία ε, πρέπει να περάσουμε από μια μακρά διαδικασία υποβολής δηλώσεων. Δηλαδή πολλές διατυπώσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα, θα διευκολύνουμε όσους ε, δραστηριοποιούνται στον τομέα. Τον Οκτώβριο του 2010 ε, υλοποιήθηκε η προηγούμενη οδηγία και θέλουμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες στον τομέα της ναυτιλίας. Θέλαμε τότε, το 2010, αλλά τελικά δεν το πετύχαμε γιατί οι ε, η υποβολή δηλώσεων ε, έχει πολλές ε, διαφορές από κράτος σε κράτος. Η νέα πρόταση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη εναρμόνισης, λοιπόν, συνδυάζοντας όλες τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων σε, ένα σε μια εναρμονισμένη δέσμη και γι' αυτό δεν θέλουμε να έχουμε υπερβολικό άχθος στους επιχειρηματίες. Γι' αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιούμε τα νέα διεθνή πρότυπα και την ενιαία ε, ναυτιλιακή θηρίδα. Καλωσορίζουμε το σχέδιο πρόταση Κομισιόν. Νομίζω ότι κάνει μια προσπάθεια για να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα της παλιάς οδηγίας του 10 και η πρώτη, το πρώτο βήμα είναι η εναρμόνιση των δεδομένων. Ε, για να αντιμετωπίσουμε και το βάρος των ε, επιχειρήσεων. Ε, το σχέδιο που συζητάμε σήμερα έχει δημοσιευθεί. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα ίδια στοιχεία υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε αρχή που ελιμενίζεται το πλοίο. Και λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις του IMO για μέγιστη προσθέμενη αξία και εφαρμόζεται Χωρί επιπλέον κόστος, ε, θα πρέπει, βεβαίως γι' αυτό, οι εθνικέ αρχές να συνεργαστούν. Θα πρέπει να έχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών, τόσο να πετύχουμε την ευελιξία. Ε, όταν τα κράτη-μέλη θέλουν περαιτέρω πληροφορίε, θα πρέπει να προσέξουν τόσο ώστε να μην αυξηθεί το διοικητικό άχθο για του επιχειρηματίε. Μια ξεκάθαρη διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά ε, την λειτουργία των εθνικών θηρίδων, θα πρέπει οι αρμόδιε αρχέ να επικοινωνούν οι εθνικές και οι αυτή της ευρωπαϊκής θηρίδας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε σωστή εφαρμογή των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων που θα γίνονται άπαξ. Θέλω τα κράτη-μέλη από κοινού αν το επιθυμούν να αναπτύξουν την ενιαία θηρίδα. Αυτά βασικά είναι κάποια από τα βασικά θέματα της έκθεσης και τώρα είμαι ανοιχτή για τροπολογίες. Έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές, ε, οι σκιώδεις συγητές ε, και εγώ και με την Κομισιόν επίσης έχουμε συζητήσει και είμαστε στη φάση συζήτησης και τροπολογιών. Είναι νομίζω όμως πολύ σημαντικό αυτό για τον ευθυλιακό τομέα. Ειδικά αν θέλουμε να αναπτύξουμε εμπορικού δεσμούς με τον υπόλοιπο κόσμο και εντός της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να γίνει και είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ κύριε Κλούν. Από του σοσιαλιστές, η κυρία Άντερσον. Um, Knut can't be here, so I'm not going to say very... Δεν θα μακρηγορήσω. Ε, θα μιλήσω στο όνομα συναδέρφου που επικροτεί τις εργασίες ε, της εισηγήτριας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόταση αυτή. Στηρίζουμε τον στόχο της ενίας θηρίδας καθώς και την μείωση του γραφειοκρατικού άχθους. Είναι σημαντικό η νομοθεσία να μην αποδυναμώσει την ε, εποπτεία και είμαι βέβαιος ότι η συγκίτρια θα το λάβει αυτό υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας καθησυχάσει όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών στο παράρτημα. Γενικά πάντως ε, προσλέπουμε στη συνέχιση των εργασιών πάνω στην πρόταση αυτή. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ θετική. Ευχαριστούμε κύριε Άντερσον. Ε, κυρία Μάισνερ. Ναι, σας ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, δεν ε, μπόρεσα να ακούσω αυτά που είπε η συγγήτρια. Ε, με δυσκολεύει πολύ όταν τροποποιείται η ημερήσια διάταξη. Ήμουνα σε άλλη επιτροπή. Πάντως γνωρίζω ότι περιέχεται στην έκθεση αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ενιαίας θηρίδας. Έπρεπε να το έχουμε κάνει πριν από πολύ καιρό. Οι εθνικές ενιαίες θηρίδες είτε δεν έχουν εφαρμοστεί είτε έχουν εφαρμοστεί με πολύ κατακαιρματισμένο τρόπο ε, στη Γερμανία, για παράδειγμα. Οι προτάσεις στην έκθεση είναι πολύ καλές. Ε, υποθέτω ότι στις τροπολογίες μας ε, θα θέλουμε να εξετάσουμε τα κράτη όπου λειτουργεί καλά η ενιαία θηρίδα και ελπίζουμε εκεί να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν οι εθνικές ενιαίες θηρίδες. Προσβλέπω στη συνέχιση της ε, συνεργασίας διότι νομίζω ότι έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, μεταφορά εμπορευμάτων. Είναι πάντα θετική η χρήση ψηφιακών μέσων για να έχουμε πιο αποτελεσματικές μεταφορές. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μάισνερ. Και να λάβω το λόγο και εγώ ως κοιόδηση Κυρία Κλούν, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για το πολύ αξιόλογο έργο σας. Γιατί έχουμε όλοι κοινό στόχο. Το στόχο που υπερασπίζεται και το κείμενο. Είναι και επιτέλους η ώρα να εναρμονίσουμε τις διοικητικές διαδικασίες εισόδου και εξόδου ελιμενισμού και απόπλου των σκαφών από τις ευρωπαϊκούς λιμένες. Και αυτός είναι βασικός στόχος μας και κυρίως να μειώσουμε τα φαινόμενα θέμη του ανταγωνισμού μεταξύ των οδικών και των αυτιλιακών μεταφορών. Γιατί αυτό είναι σημαντικό διακύβευμα που λαμβάνουμε υπόψη στην Επιτροπή Μεταφορών. Στην Ευρώπη ένα φορτηγό μπορεί να περάσει τα σύνορα χωρίς κανένα πρόβλημα. Ενώ στις ναυτιλιακές μεταφορές ένα πλοίο που ελιμενίζεται πρέπει να αναλάβει πολύ ε, βαριές διοικητικές διατυπώσεις με τεράστιο κόστος δυσβάσταχτο. Επίσης, αυτό επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών, που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες και διατυπώσεις. Η κυρία Κλούν με την έκθεσή της ε, ακολουθεί το σωστό δρόμο και ελπίζω να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι σε κάποια ζητήματα που αναφέρατε, δηλαδή το θέμα της εναρμόνισης των δεδομένων ε, ήρθε η ώρα να εναρμονίσουμε και τα δεδομένα. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Επίσης, ε, τεχνολογική ουδετερότητα και αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει. Και επίσης να, ε, να παρακολουθήσουμε το έργο και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για αυτά τα τρία σκέλη που μας ενδιαφέρουν. Και γι' αυτό θα προσπαθήσω να εμπλουτίσω με τροπολογία στο κείμενό σας που είναι προς σωστή κατεύθυνση. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Κοσένσκα εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης ΜΟΥΒ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω να μην χτυπήσετε πολύ άσχημα στο πόδι. Δεν πρέπει να βιάζετε και να τρέχετε και αν χτυπήσατε φροντίστε το πόδι σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ε, έσπασα το πόδι μου όχι ερχόμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν προηγούμενο το ατύχημα. Ε, προσπάθησα να έρθω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ε, πραγματικά έχω διαβάσει την έκθεση και ελπίζω ότι στις συναντήσεις που έχουν οι συνάδελφοι και που είχαν πριν από δύο εβδομάδες με τους και ηγητές σας χρησιμεύσαν για να διαλευκανθεί περαιτέρω η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν χρειαστούν και ακόμη νέε ναι, συνεδριάσει, κανένα πρόβλημα, είμαστε στη διάθεσή σα. Επίση, να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για την έκθεση, αλλά και γενικώ για τη θετική σα αντίδραση και τη, της και των μελών της Επιτροπής σας σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της αναγκαιότητας, της επιτακτικής ανάγκης να καταλήξουμε σε πιο εναρμονισμένο και προηγμένο σύστημα για να πλουστεύσουμε την υποβολή δηλώσεων των πλοίων που ελιμενίζονται στους ευρωπαϊκούς λιμένες και εσείς κυρία Πρόεδρε και κυρία Μάισνερ πολύ εύστοχα μιλήσετε για το σημαντικό αντίκτυπο που θα έχει τέτοια απλούστευση στην διευκόλυνση των ευρωπαϊκών αυτιλιακών μεταφορών. Θα γίνουν οι ναυτιλιακές μεταφορές πιο ανταγωνιστικές και πιο εύχριστες γιατί είναι και πιο βιώσιμος τρόπος μεταφοράς. Και κάτι άλλο που δεν έχει υπογραμμιστεί αρκετά ίσως στην νομοθετική πρόταση. Πάντως όταν συντάξαμε τη μελέτη επιπτώσεων, ο αντίκτυπος ε, ε, των αλλεπάλων και περίπλοκων ε, διατυπώσεων και το κόστος και το ο φόρτος που δημιουργείται για τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους στην αυτιλία είναι πολύ σημαντικό. αυτό θα μειωθεί λοιπόν αυτός ο αντίκτυπος. Επίσης, χαιρόμαστε που αναγνωρίζετε και εσείς την επιτακτική ανάγκη για την θέσπιση μιας ενίας ναυτιλιακής θηρίδας και ελπίζω οι δύο τα δύο αρμόδια σκέλη της νομοθετικής αρχής να συμφωνήσουν και να καλύψουμε τις καθυστερήσεις μέχρι το φθινόπωρο. Είναι περίπλοκο το θέμα, πάντως και με την δική σας δέσμευση αλλά και με την προθυμία της Προεδρίας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ποιο είναι το υπόβαθρο αυτής της πρότασης Εσεί στις τροπολογίες σας προτείνετε να μην έχουμε μια νέα ημερομηνία, μια νέα προθεσμία από τη στιγμή που συμφωνηθεί μια προθεσμία στο σύστημα. Συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Σε ό,τι αφορά τι διευκρινήσεις επίσης για την επικοινωνία μεταξύ των ε, παρόχων δεδομένων και των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να είναι αφίδρομη η επικοινωνία διασαφιστών και αρμόδιων αρχών. Επίσης, θα πρέπει η πρόταση να είναι φιλική προς το χρήστη, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και των εφοπλιστών και των πλειοκτητών, να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο υποβολής δηλώσεων και εναρμονισμένο και για τις ναυτιλιακές αρχές και για τις πολυτροπικές αρχές. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για να διευκολυνθεί η μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η βασική μας κατεύθυνση. Επίσης θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς τις προσδοκίες που μπορεί να έχουμε από τις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές αρχές από τη στιγμή που θα μπουν τα δεδομένα στο σύστημα. Για παράδειγμα, ε, προθεσμία για την ε, έγκριση των προτάσεων ή την κύρωση των προτάσεων, επικύρωση των προτάσεων ή επίσης η οργάνωση θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο και για τις αρμόδιες αρχές και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, όπως είπατε και σήμερα, ε, έχουμε εθνικές ενιαίες ε, θηρίδες που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα ενιαίας ναυτιλιακής θηρίδας. Μόνο έτσι θα διευκολύνουμε τις ναυτιλιακές μεταφορές και θα απλουστεύσουμε τις διοικητικές διατυπώσεις για τον ρελιμερισμό. Και ε, ακόμη και αν υπάρχουν και παραμείνουν κάποια εναλλακτικά συστήματα θα πρέπει να υποκαταστήσουν αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον ενιαίας ναυτιλιακής θηρίδας που είναι ο απότερος σκοπός μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές και από τις τροπολογίες. Ευχαριστώ και προσβλέπουμε σε συνέχιση της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ και καλή ανάρρωση για το πόδι σας. Ακούσατε τι σας είπα από τη μετάφραση. Και φροντίστε το πόδι σας. Αυτό σας είπα. Μιλήσατε για την ενίσχυση της, των πολύτροπων μεταφορών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στον 21ο τομέα. Ε, συγγνώμη, αιώνα. Η κυρία Φώστερ μόλις ήρθε, θα της δώσω το λόγο για να κάνει τις παρατηρήσεις της, μια και είναι η συγγήτρια εδώ και μια και είστε σκιώδης η συγγήτρια, καλό να σας δώσω το λόγο. Κυρία Φώστερ, έχετε τον λόγο. Yeah. Which report are Για ποια έκθεση μιλάμε? Κλάμε. Συγγνώμη, ναι, κατάλαβα ότι τροποποιήθηκα, τροποποιήθηκε η ημερήσια διάταξη. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλάει για την ενιαία θηρίδα. Βρισκόμαστε στην αρχή τη συζήτηση αυτή. Α, όχι, δεν θα σχολιάσω, διότι δεν μπόρεσα να ακούσω όλε τι παρατηρήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Ε, ε, θα συνεννοηθούμε. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. I really wanted to. Η δική μου έκθεση ακυρώθηκε από ό,τι κατάλαβα. That's all right, only around 3,000 miles an hour for Maya. Décidément. Eh ben, décidément, il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement pour le rapport de Madame, de Monsieur Mayer et Monsieur. Ήρθατε για την έκθεση Mayer ε, και τελικά ο κύριος Μάιερ δεν είναι εδώ και θα τη συζητήσουμε αυτή την έκθεση. Η έκθεση αυτή θα συζητηθεί όμως την επόμενη φορά. Κυρία Κλούν, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους και όλους τους για τα σχόλιά τους. Βλέπετε ότι υπάρχει αρκετή συνετική διάθεση για αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν δυσκολίες τελικά. Έχουμε συμφωνήσει με την Κομισιόν να έρθουν στην, στο Στρασβούργο σε δύο εβδομάδες για να μας διευκολύνουν ε, για το θέμα μας και εκεί θα ρυθμίσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Είναι κατεπήγον το θέμα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ στην ε, Επιτροπή προσπαθούμε να, να είμαστε σε επαφή με τους σκιώδεις συζητητές και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την ε, καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες και για την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Θα είμαι στη διάθεσή σας για να δω ότι θα, τη διάθεση υπάρχει από τους άλλους. Ε, κοιτάξτε, δεν νομίζω θα υπάρχει πρόβλημα, μια και υπάρχει σοβαρή συνένεση, η οποία θα μας διευκολύνει. Μιλήσατε για μια αρέωση, για μια αποδυνάμωση της πρότασης της Κομισιόν. Δεν είναι καθόλου αυτή η πρόθεση. Ε, το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Και δεν θέλουμε διάφορε χώρε να ζητάνε το ίδιο πράγμα, ε, σε διάφορα λιμάνια δηλαδή, να ζητάνε το ίδιο πράγμα από το ίδιο πλοίο. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Εναρμόνιση θέλουμε, όχι αποδυνάμωση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και του σκιώδη συζητητέ για τη συζήτηση, η οποία ε, ήταν πολύ καλή και οι σκιώδη συζητητέ έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συζήτηση. Η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι 20 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Και τώρα θα ζητήσω από όλου όσου δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην αίθουσα να βγουν παρακαλώ γιατί θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας και κλεισμένων των θυρών για να ενημερωθούμε για τους τριμερείς διαλόγους και σας ζητώ λοιπόν όλους εσάς που δεν πρέπει να είστε στην αίθουσα να βγείτε τώρα και γρήγορα μάλιστα. Θα ήθελα επίσης το web streaming να σταματήσει.